Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Έτσι θεωρείται ότι κυρώνονται τα πρακτικά αυτά. Από την ομάδα έχω διορισμούς σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο